Ε, μέσω της ε, κοινή ε, συνεργασίας, κοινής επιτροπής συνεργασίας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ κύριε Επίτροπε. Τελειώνει εδώ πέρα η συζήτηση για το Αζερβαϊτζάν. Η συζήτηση θα γίνει μετά το τέλος του επόμενου θέματος που είναι η Λευκορωσία. A první na řadě, kdo vystoupí, je pan poslanec Maštálka, prosím. Maštálka είναι ο πρώτος ομιλητή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ενώ προσπαθούμε να αξιολογούμε αντικειμενικά τις εγχώριες ε, καταστάσεις, ε, οι εταίροι μας προσπαθούν να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Θα ήθελα να σας πω ως γιατρός ότι η βία από όπου και αν προέρχεται είναι βία και είναι αντίθετη με τις κοινέ μας αρχές και αξίες. Αυτοί οι οποίοι είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή θα πρέπει να χαίρουν συνθήκων υγείας ε, ε, αξιοπρεπών και παρκών και ανθρώπινης μεταχείρισης. Με τη Λευκορωσία δεν είναι δυνατόν η στόχη της συνεργασίας να είναι εφικτή λόγω των μέτρων που έχει λάβει η χώρα αυτή. Η δήλωση της Πράγας παραβιάζεται και καθυστερούν οι αλλαγές που θα βοηθήσουν την αμοιβαία συνεργασία. Οι για τη δημιουργία μιας ενιαίας Ευρώπης είναι κάτι που είναι πολύ προσφυλές, ιδίως για τους νέους στη Λευκορωσία. Θα πρέπει να θεωρήσουμε την απόψή μας και να ξανασκεφτούμε κατά πόσον οι περιορισμοί είναι το κατάλληλο εργαλείο Θέλουμε η κοινότητα των πολιτών της Λευκορωσίας να μας ω ένα πραγματικό φίλο. Έχουμε την 25η επέτειο από την καταστροφή του Τσέρνομπιλ. Θα ήθελα να παρακαλέσω να δούμε κάπως διαφορετικά τη Λευκορωσία, να τη δούμε ως ένα κράτος που έχει υποφέρει τα μάλα. Είναι μια καταστροφή αυτή του Τσέρνομπιλ που έπληξε τη Λευκορωσία, το λαό της και δεν τους επέτρεψε να συμμετάσχουν στην επίσημη τις επίσημες τελετές. Τώρα, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι που είπε ο κύριος Τάνοκ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μιλά κανεί γρήγορα αγγλικά. Μ' αρέσουν τα αγγλικά. Είναι η γλώσσα του Σέξπιρ. Ίσως ε, καλό θα ήταν να προσπαθήσετε να μιλήσετε γρήγορα στη χώρα του Γκέτε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ κύριο Παλέτσκης. Thank ε, Σας ευχαριστώ. Τους τελευταίους πέντε μήνες από τις 19 Δεκεμβρίου και μετά η πολιτική κατάσταση στην Λευκορωσία όλο ένα και υποβαθμίζεται. Επιδεινώνεται εκφοβισμό, εκφοβισμός, η άσκηση πίεσης και απειλών, η δίωξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στην Λευκορωσία παραβιάζονται όλες οι διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο διάλογος ολοένα και δυσχεραίνεται. Από το Μίνσκ έχουμε πολλές ε, κατηγορίες ε, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαπολύονται κατηγορίες ενώ εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών. Η αντιπολίτευση θεωρούμε ότι βρίσκεται στο, στο πλευρό της κοινωνίας των πολιτών εδώ θα μπορούσε να μας συνδράμε και το Κίεβο, η Ουκρανία στον διάλογο για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Σας ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής ο κ. Πρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην προηγούμενη παρέμβαση όπως και άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκα στην συνεδρίαση της συνοβουλευτικής διάσκεψης του Euronest που έγινε απουσία βουλευτών της Λευκορωσίας γιατί ε, δεν εκλέγονται δίκαια και ελεύθερα οι βουλευτές στο Μίνσκ. Επιπλέον η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κρίσιμη. Όλοι εξηγηθήκαμε μετά τα όσα έγιναν με βάρος των διαδηλωτών ε, ε, τον Δεκέμβριο. Έξι ανθυποψήφοι του κυρίου Λουκασέγκα είναι ακόμη φυλακισμένοι και υπόδικοι. Το ίδιο και τα επιτελεία τους μόνο και μόνο για τη συμμετοχή τους. Θεωρώ πως υπάρχουν δύο σημαντικές πτυχές. Πρώτον, χρειάζεται μία ανεξάρτητη έρευνα. Δεύτερον, πρέπει να επεκταθούν οι οικονομικές κυρώσεις και σε κρατικές εταιρείε που παίζουν σημαντικό ρόλο στο καθεστώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Όγιουλαντ κατόπιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε την κατάσταση της Λευκορωσία για τέταρτη φορά φέτος όμως. Οι πολιτικοί κρατούμενοι που συνελήφθησαν το Δεκέμβριο ακόμα δεν έχουν ελευθερωθεί. Είμαστε ευγνώμονες στο Συμβούλιο για το ότι επανεισήγαγε κυρώσεις για την Βίζα και πάγωμα των παρουσιακών στοιχείων των Λευκορώσων αξιωματούχων που δείχνουν την ανησυχία μας για το λαό της Λευκορωσίας και ότι αυτά δεν είναι μόνο λόγια. Ίσως δεν ήμασταν αρκετά σαφείς. Γι' αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει περιοριστικά μέτρα ε, εις βάρος το καθεστώτος Λούκασέγκα στοχευμένες κυρώσεις κατά κρατικών επιχειρήσεων θα έχουν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορούν να αγνοήσουν οι αρχές της Λευκορωσίας. Το εγκληματικό καθεστώς Λουκασένκο βασίζεται κυρίως στην εξαγωγή χημικών βαριάς βιομηχανίας και υφασμάτων. Αποκόπτοντάς τους από την ευρωπαϊκή αγορά δείχνουμε την αποφασιστικότητά μας να ανατρέψουμε το καθεστώς Λουκασένκα είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας το να κάνουμε τη διαφορά. Χρειάζεται αλλαγή του καθιστώτος για τον λαό της Λευκορωσίας. Δεν πρέπει να του αρνούμαστε την ελευθερία. Ευχαριστώ. Κυρία Ογιουλάντ. Κύριος Καμίνσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για πολιτική, για ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της κατάστασης της, της Θα ήθελα να το δω λίγο ασύμβατα το θέμα, όχι συμβατικά μάλλον, και να σας θυμίσω δύο ονόματα που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Το πρώτο είναι ένας φίλος μου, Νατάλη Λιμπίτσκο, που πρόσφατα μόλις απελευθερώθηκε από την φυλακή, μετά από πάνω από 100 ημέρες ε, όπου κρατεί δεν ήταν δικαιολογημένο αυτό από νομική πλευρά κατά την άποψή μου και θα ήθελα να του στείλουμε ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης. Γιατί πραγματικά αξίζει την στήριξή μας. Επίσης ε, κάτι άλλο είναι ο ένα άλλο όνομα, ο Αντρέ Ποτσόνον από την Πολωνία, ένας ανεξάρτητος ε, δημοσιογράφος που κρατείται στη φυλακή, που διώχθηκε επειδή ο Λουκασέγκο και το καθεστώς του φοβάται την ελευθερία λόγου. Μια ελευθερία που είναι η βάση της δημοκρατίας. Εμείς ως δημοκράτες θα πρέπει να πούμε ναι στην ελεύθερη Λευκορωσία, ναι στη δημοκρατία στη Λευκορωσία, ναι στους Λευκορώσους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Mr. Romeva Irueda ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα. Κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμη φορά λυπούμε που υπάρχει αυτό το καθεστώς εκφοβισμού και καταστολής στη Λευκορωσία, τις συνεχιζόμενες παρενοχλήσεις και διώξεις σημαντικών προσωπικότητων της αντιπολίτευσης, όπως είναι το Δεκέμβριο του 2010. Δεύτερον, καταδικάζω στενάρα τις ε, δίκες ε, που έγιναν ε, για μαζικές ταραχές δεν στηρίζονται από το διεθνές δίκαιο. Έγιναν οι δίκες πίσω από κλειστέ πόρτες, δεν υπήρξαν σωστές συνθήκες, ούτε καν σε κάποιες περιπτώσεις υπεράσπιση δεν είχαν οι κατηγορούμενοι. όσοι προσπάθησαν να τους υπεστηρίξουν ε, μέχρι που έχασαν και τη θέση τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τέλος, θέλω να ε, εκφράσω τη λύπη μου που δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Θέλω να ζητήσω την ανεφόρον απελευθέρωση όσων διαδηλωτών είναι στη φυλακή. Και πρέπει να πέσουν όλες οι κατηγορίες σε βάρος τους. Ευχαριστώ οι ομιλητέ εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Προτάσεβιτ για το ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Πράγματι, η κατάσταση στη Λευκορωσία επιδεινώνεται καθημερινά. Και στο πολιτικό και στο οικονομικό του σκηνικό. Ε, από πολιτική άποψη και σε ό,τι αφορά τι ελευθερίε των πολιτών, βλέπουμε δίκες τελείως παράλογες κατά των άλλων υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές. Η σύλληψη του δημοσιογράφου ήδη αναφέρθηκε, αλλά και από οικονομικής άποψης, η υποτίμηση σε σχέση με το ρούβλι ε, και οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ο Λουκασέγκο χάνει τον έλεγχο όχι μόνο εκτός χώρας, αλλά και σε όχι μόνο μάλλον στο εσωτερικό τη χώρα, αλλά και σε το διεθνέ προσκήνιο με τι κατηγορίε του κατά του κυρίου Μπαρόζο και το καθεξή. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να περάσουμε και να αναλάβουμε δράση με το άρθρο 8 του, όπω ε, αναφέρει και το ψήφισμά μα. Ε, ε, θα πρέπει να μιλήσουμε μια γλώσσα από ο κ. Λουκασέγκο να μπορεί να την καταλάβει με οικονομικέ κυρώσει, ώστε να σταματήσει η καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτέ οι παράλογε δίκε να πάυσουν. Αυτή είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ο κ. Λουκασέγκο και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να οδεύσουμε. Σα ευχαριστούμε κύριε Προτάσεβιτ, ο κ. Ρέπο, εκ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Μπορούμε εδώ να μιλήσουμε για την τελευταία δικτατορία στην Ευρώπη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τα πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Οι τελευταίες προεδρικές εκλογές δεν ήταν δημοκρατικές. Δεν υπήρξε καμία ελευθερία έκφρασης ούτε συγκέντρωσης. Τα μέλη της αντιπολίτευσης, τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών έπεσαν θύματα παρενόχλησης του, αν μη τι άλλο. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας ε, να συμμετάσχει ενεργά στον πολιτικό διάλογο όλοι οι πολίτε τη χώρα. Διότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, θεμελιώδη ελευθερίε είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα αποσιωπούμε. Θα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Θα πρέπει η Λευκορωσία να βελτιώσει την κατάστασή τη σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι καθαριστικό αυτό στα πλαίσια τη πολιτική γειτονία μα και τη πολιτική συνεργασία προ Ανατολά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν λύσει για την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ κύριο Ντόνσκι για του φιλελεύθερου και δημοκράτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει ένδειξη για το ότι μπορεί να αλλάξει από μόνο του το καθεστώ Λευκορωσίας Οπότε νομίζω πως μόνο υπό ισχυρή πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να αναμένουμε να γίνει κάτι. Παραβιάζονται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες και βλέπουμε πως οι αρχές Λευκορωσίας τον τελευταίο μήνα έδειξαν την περιφρόνησή τους για θεμελιώδη δικαιώματα όπως το δικαίωμα του συνέρχεστε και η ελευθερία έκφρασης. Εδώ πέρα μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς δεν αλλάζει ο Λουκασένκο και το καθεστώς του. Αλλά δεν μπορούμε να τελειώσουμε έτσι απεσιόδοξα. Πρέπει να αντιληφθούμε πως πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στους Λευκορώσους πως είναι ευπρόσδεκτοι στην Ευρώπη. Και νομίζω καλό ήταν να μιλήσουμε για τις αρχές μας λόγω των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μην παρασυρώμαστε από το ότι προσπαθεί να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκνευρίσει προσωρινά τη Ρωσία και αντιστρόφως. Πρέπει να αξιολογηθεί με βάση αρχές η Λευκορωσία και να ασκήσουμε καλύτερη πίεση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Ντόνσκης. Κύριος Πορέμπα για τους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά μέσο όρο κάθε δύο μήνες από την αρχή του έτους μιλάμε στην Ολομέλεια για το τι γίνεται στη Λευκορωσία. Νέε περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νέα ονόματα ηγετών τη αντιπολίτευση που καταλήγουν στη φυλακή που δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για ΜΚΟ και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Πράγματι θα πρέπει να καταδικάζουμε τέτοιες δραστηριότητες, αλλά θεωρώ πως είναι εξίσου σημαντικό, αν όχι πιο σημαντικό για εμάς, να εμπλακούμε στην οικοδόμηση της ε, κοινωνίας των πολιτών και στο να στηρίξουμε ΜΚΟ και ελεύθερα ΜΜΕ. Στη Λευκορωσία επίσης όσον αφορά τις οικονομικές κυρώσεις φαίνεται πως έχει φτάσει η στιγμή να τα εφαρμόσουμε αυτά. Σήμερα θα ψηφίσουμε το ψήφισμα που στόχο έχει να δώσει ηθική στήριξη στην κοινωνία της Λευκορωσίας. Θεωρώ πως θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα μέτρα ή οικονομικά κυρώσεις που θα αποκαταστήσουν τη δημοκρατία στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία, Η κυρία Μορβά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το θέμα της συζήτησής μας Έχω και εγώ μία ερώτηση. Τι θα λέγατε εάν ένα μέλος της κυβέρνησης Λουκασένκο βρισκόταν σε ένα-δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γινόταν πρόεδρος της Επιτροπής Ελευθεριών. Τι θα λέγατε τότε και πότε θα φτάσουμε στις ε, συζητήσεις μας ε, στο σημείο το απόγευμα της πέμπτης σε αυτό το σημείο. Έχω λοιπόν ε, ένα λεπτό. Εγώ έθεσα το πρώτο ερώτημα όσον αφορά τα μέλη της κυβέρνησης Λούκασέγκο. Έχουμε και τον Ούγκρο Λουκασένκο και ένα μέλος αυτής της κυβέρνησης, ο βουλευτής King Γκέντς, είναι αναπληρωτής πρόεδρος Επιτροπής Ελευθεριών και είναι και συμβουλές. Πώς ανεχόμαστε τον Ούγκρο Λουκασένκο και γιατί ακριβώς ε, δεν είναι τόσο γνωστός. και ακριβώς όπως και ακριβώς τα ίδια προβλήματα επέδειξε. και απευθύνουμε έκκληση άρα να συμπεριφερθεί σωστά η κυβέρνηση Λευκορωσίας αλλά τι κάνει και τι έκανε και η Ουγγαρία παντού καταπνίγονται και στις δύο χώρες ε, με βία οι διαδηλώσει Εμένα με αποζημίωσαν γιατί μου έριξαν κρυγόνο στα μάτια. Άνθρωποι στην Ουγγαρία είναι στις φυλακές, ε, μιλάμε για ηγετικές προσωπικότητες που κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις ε, και έπαιξαν ένα ρόλο. Στις ΗΠΑ εξακολουθεί να υπάρχει εντωμεταξύ η θανατική ποινή και στον Κουαντανάμο να υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, καταδικαστές ε, μέθοδοι που χρησιμοποιεί επίσης η κυβέρνηση Λουκασέγκο. Állami Και εσείς θέλετε κυρώσεις κατά της κυβέρνησης Λουκασέγκο. Και σβήνει το μικρόφωνο. Κατόπιν ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, δεν συμφωνώ πάντα με τη συνάδελφο Μάστα, αλλά σήμερα συμβαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω πως όλα τα κόμματα πρέπει να αγωνιστούν για να έρθει επιτέλους η δημοκρατία στην ε, Λευκορωσία. Και δεύτερον, να μιλήσω υπέρ της πολυγλωσσίας. Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι από μία χώρα, προερχόμουν από μια αυτοκρατορία των Αψβούργων η οποία κατέρευσε γιατί κατέληξε να φύγει από μέσα η μεγαλύτερη κοινότητα της η γερμανόφωνη. Είμαστε λοιπόν ε, υπέρ της πολυγλωσσίας για μικρές και μεγάλες γλώσσες. Τώρα όσον αφορά την ε, Λευκορωσία. Πριν από 20 χρόνια ελευθερώθηκε η Κροατία και η Σλοβενία. Και ήμουν εκεί. Και Αύγουστο του ίδιου έτους Ουκρανία και Λευκορωσία και κανείς δεν σκεφτόταν πως μετά από 20 χρόνια θα υπήρχαν ακόμα δικτατορίες στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχουν, υπάρχει η Λευκορωσία, υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις στην Ρωσία, οπισθοχωρήσεις στην Ουκρανία, προβλήματα στη Μολδαβία και υπερδνηστερία και πρέπει να ομολογήσουμε πως υπάρχει κίνδυνος για την ελευθερία σε ολόκληρη την ανατολική γειτονιά μας. Οπότε Πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα αυτά, να σκεφτούμε στρατηγικά και να γίνει η ελευθερία μέτρο των σχέσεών μας με την ανατολική μας γειτονιά. Και όχι μόνο κατά της Λευκορωσίας. Ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ, κύριο Σμιγκάλσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς ε, κάτι προσωπικό. Μία οργάνωση ε, που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ήρθε σε επαφή μαζί μου και ζήτησε να παρασχεθεί προστασία σε έναν από τους αντικαταστατικούς που κρατείται σε φυλακές, ο κύριος Πανταρένκο συγκεκριμένα. Όσους σας ενδιαφέρει το θέμα αυτό, θα ήθελα να το έχετε υπόψη σας. Είναι σημαντικό προσωπικά και εμείς να παρέχουμε προστασία σε άτομα τα οποία κρατούνται στις φυλακές. Νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορούμε προσωπικά να κάνουμε για όλα ε, τα άτομα τα οποία κρατούνται στις φυλακές της Λευκορωσίας. Ζητούμε για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει βέβαια να έχουν τη μορφή κυρώσεων γιατί αυτή είναι η μόνη, η μόνη γλώσσα που θα καταλάβει ο Λουκασέγκο καταλαβαίνει τη γνώσα των επιχειρήσεων και τη γλώσσα της εξουσίας. Για να σωθεί η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα που καταλαβαίνει το Μίνσκ. Έχει ξαναυποθεί στην ε, Ολομέλεια, αλλά δεν έχουν τα λόγια συνοδευτεί από τις απαραίτητες πράξεις. Όλοι μας όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να μιλούν για αυτό το θέμα. Θα πρέπει όμως και εμείς να μιλούμε στις χώρες μας, ε, στις κυβερνήσεις μας, γιατί και οι κυβερνήσεις μας μπορούν να προσπαθήσουν να πείσουν τον κύριο Λουκασέγκο να εγκαθιδρύσει τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Κυρία Κόρχολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Λουκασέγκο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, επανεκλέγει, επανεξελέγει μάλλον. Αλλά ξέρουμε ακριβώς πώς διεξήχθησαν αυτές οι εκλογές. Ξέρουμε ότι ήταν οθευμένες και ότι φημώθηκε η αντιπολίτευση. Εκατοντάδε φυλακίστηκαν με, την, το πρόσχημα ότι υποκίνησαν διαμαρτυρίε και διαδηλώσει. Ο πρόεδρος έχει στα χέρια του συγκεντρωμένη όλη την εξουσία. Μιλάμε για ένα απολυταρχικό καθεστώ. Καταλάβαμε ότι οι πρώτες προσπάθειες εκδημοκρατισμού κατεπνίγησαν. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς από τη δική μας πλευρά να γίνουμε αστηρότεροι. Θα πρέπει να επιμείνουμε για όσου αθλητικέ οργανώσει έχουν σκοπό να οργανώσουν ε, κάποια γεγονότα στη χώρα αυτή τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να τι αποθαρρύνουμε. Σα ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διεθνή κοινότητα, εντό τη οποία βέβαια λειτουργεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλεί τι λευκορωσικέ αρχέ να σεβαστούν επιτέλου τι υποχρεώσει του. Να πάυσουν την ε, καταπίεση της αντιπολίτευσης, να απελευθερώσουν τους αντιφρονούντες που έχουν ε, συλληφθεί, να πάυσουν τα μέτρα καταπίεσης και θύμωσης του τύπου, των κοινωνίες των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να είναι δίκαια και διαφανής. Οι αρχές της Λευκορωσίας θα πρέπει να κατανοήσουν ότι χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου, χωρίς Μάλλον και σύμφωνα με, την, με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου αφορμή τη Σύνοδο Μα συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρο, δυσκολεύονται οι Γερμανοί να παρακολουθήσουν το ρυθμό σα. Ε, οι αρχέ τη Λευκορωσία θα πρέπει να καταλάβουν ότι χωρί το σεβασμό των θεμελιδών ε, ελευθεριών και του κράτου δικαίου και σύμφωνα με την κοινή δήλωση στη Σύνοδο κορυφή για την ε, πολιτική συνεργασία τη Ανατολά ε, τον Μάιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κάνει πλέον καμία δράση στήριξη τη Λευκορωσία. Ευχαριστούμε, κύριε Λουνάτσεκ. Η κυρία Λουνάτσεκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα τον λόγο γιατί ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Μορβάη. Η King Against δεν είναι από το κόμμα μου. Αλλά δεν μου αρέσει το πώς χρησιμοποιήσατε μια συζήτηση για την τελευταία δικτατορία στην Ευρώπη του κυρίου Λουκασέγκο για να δυσφημίσετε ένα έντιμο μέλος του Κοινοβουλίου και να την πείτε Ούγκρο Λουκασέγκο. Δεν συμφωνεί αυτό με τις αξίες που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο όλοι έχουμε εκλεγεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόρβαϊ έχει μια μπλε κάρτα. Ναι, αναρωτιέμαι. Με ακούγατε όταν έλεγα πως είναι μέλος της ε, ουγγρικής κυβέρνησης ε, Λουκασέγκο, του κυρίου Ντούνσον. Απαντήστε μου, τι ξέρετε. Τι ξέρετε για τις μαζικές παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία το 2006. Συνοψίστε τα. Δεν ήταν λιγότερο σοβαρές σε σοβαρότα και αριθμό από αυτές του Λουκασέγκο και ως δικηγόρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζω και τις δύο περιπτώσεις. Οι σύντροφοί σας πυροβολούσαν στα μάτια τους ανθρώπους αυθαίρετες συλλήψεις ό,τι έκανε και ο Λουκασέγκο. Και οι δύο είναι απαράδεκτοι. Και εσείς ως βουλευτές πρέπει να αντιπαλέψετε και τους δύο κυρία Λούνατσεκ και ο κύριο Σούλτς. Ε, μάλλον ε, τα έχετε μπερδέψει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κόμμα Λουκασέγκο στην Ουγγαρία. Δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, δεν είμαι από την Ουγγαρία. Αλλά αρνούμε να δεχτώ μέλο του Κοινοβουλίου να ασκεί κριτική σε συνάδελφο εδώ μέσα και να λέει ότι είναι μέλο δικτατορικού κόμματο σε μια άλλη χώρα που δεν είναι μέλο κράτο. Τελεία. Κύριε Σούλτς, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Κίνγκα Γκέντς είναι μέλος ομάδας μου. Μπορούμε για τον... Μπορούμε να είμαστε υπέρ κατά του Φέρεντς Γιόρτσανη. Μπορεί να είναι υπέρ ή κατά κανείς της Κίνγκα Γκέντς. Αυτό είναι θέμα του καθενός και θέμα ελευθερίας. Και ανεξαρτήτως του εάν ε, είναι κανείς υπέρ ή κατά ενός ατόμου. Η συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ πέρα γίνεται για την τελευταία δικτατορία που υπάρχει στην Ευρώπη. Και μιλάμε για έναν αδίστακτο και αιμοσταγή δικτάτορα. Και είναι απολύτως απαράδεικτο ένα ερετό μέλος της ομάδας μου να συγκρίνεται με έναν αιμοσταγή δικτάτορα. Πρέπει να το απορρίψει το Κοινοβούλιο, ειδικά από εκπρόσωπο ενός κόμματος που δεν συμπεριφέρεται και πάρα πολύ καλά και μάλιστα συμπεριφέρεται με λόγια και πράξεις μίσους κατά της μειονότητας Ρωμά στην χώρα τους. Αυτά όσον αφορά την κυρία Κίνγκα Γκέντς. Λοιπόν, θα περάσουμε στον επόμενο μιλητή μας που είναι ο κύριος Στάνο. Κυρία Μορβάη, ζητώ συγγνώμη αλλά ε, ήδη ε, είχατε την ευκαιρία σας. Τώρα, όπως σας είπαν και οι προλέσσαντες, μιλάμε για τη Λευκορωσία. Ναι, πράγματι, εγώ θα μιλήσω για τη Λευκορωσία και όχι για την χώρα πολιτική της Ουκαρίας. Ε, κατέρευσε πριν από 20 χρόνια η Σοβιετική Αυτοκρατορία. Αλλά στη Λευκορωσία σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Συνεχίζει η καταστολή, ο Λουκασέγκο και η μυστική του αστυνομία, προκλητικά ε, χρησιμοποιούν και λέγονται KGB ε, ακόμα, KGB και χρησιμοποιούν τους ίδιους τρόπους, ίδιες μεθόδου. Φαίνεται να αρέσκονται στον να εκφοβήσουν, στο να ασκούν βία κατά των δημοκρατικών ακτιβιστών. Όπω δείχνει πολύ εύγλωτα το σημερινό ψήφισμα ο Λουκασέγκο έχει εντείνει την εκστρατεία ε, παρενόχληση, δίωξη, ε, όσων είναι αντίθετοι ε, στο σιδερένιο τρόπο με τον οποίο κυβερνά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η κατεύθυνση που ακολουθεί η Λευκορωσία, να ακολουθεί στον δρόμο της δημοκρατίας. Η Λευκορωσία πραγματικά είναι ένας ε, χαμένος ε, κρίκος, ε, ο κρίκος που λείπει, το, το κομμάτι του παζλ που λείπει από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Σας ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Ρούμπιξ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω πλήρω. την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βλέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες όχι μόνο εντός Ευρώπης αλλά και εκτός. Και θα πρέπει να ακολουθηθεί ίσως μια γενική προσέγγιση Δεν θα πρέπει να κατηγορείται κάποιο μέλος μιας κυβέρνησης για κλίματα τα οποία δεν έχει διαπράξει. Υπάρχουν, υπάρχουν αντιφροντές οι οποίοι κράτονται στις φυλακές. Ε, γίνεται λόγος για δικτατορικές ε, πρακτικές. Αλλά πρέπει να δούμε τελικά τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Αν έχουν γίνει όλα σωστά και άγια. Πρέπει να είμαστε ανεκτικοί, αλλά πρέπει να υπάρχουν τα ίδια μέτρα και τα δύο σταθμά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μιγκάλσκι είχε ήδη το λόγο. Συγγνώμη κύριε Μιγκάλσκι, δεν μπορώ να σας ξαναδώσω το λόγο. Πρέπει να λήξει η συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Άντορ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί βαθύτατα για την κατάσταση στην ε, Λευκορωσία και ιδιαίτερα με τις εξελίξεις ε, μετά την παραβίαση των εκλογικών προτύπων στις 19 Δεκεμβρίου του 2010, τις δηλαδή που έγιναν οι προεδρικές εκλογές. Έχει ενταθεί η καταστολή, υπάρχουν δίκες εξέλιξη αυτόν τον καιρό κατά ε, υποψηφίων για την Προεδρία, αλλά και των υπόλοιπων ακτιβιστών που κράτονται στις φυλακές. Επίσης υπάρχουν διαδικασίες και δίκες που ίσως οδηγήσουν στο κλείσιμο δύο από τις εναπομένουσες εφημερίδες που θεωρούνται ανεξάρτητες, την Ναρόδια Βόλια και την Άσα Νίβα. Συνεχίζεται η καταστολή της ανεξάρτητης ελευθεροτυπίας. Η είπατε πρόσωπος Βαρόνια τον έχει προβεί σε γενικές και ειδικές δηλώσεις σε σχέση με τη Λευκορωσία. Έχουμε ξεκάθαρα και απερίφραστα καταδικάσει την κατάσταση στη Λευκορωσία και έχουμε απαλληλμένως καλέσει τη Λευκορωσία να θέσει ένα τέρμα στη συνεχιζόμενη καταστολή της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε ζητήσει την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και να σταματήσουν οι δίκες πολιτικών κρατουμένων και έχουμε εκφράσει βαθιές ανησυχίες μετά από καταγγελίες για βασανισμούς και άλλη κακομεταχείριση, κακοποίηση, εκφοβισμό και διάφορες άλλες ε, καστικές ατασταλίες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω επίσης ότι τον Ιανουάριο το Συμβούλιο ενέκρινε περιοριστικά μέτρα μεταξύ αυτών απαγόρευση μετακίνησης πάγων περιουσιακών στοιχείων. 175 άτομα περιλαμβάνει ο κατάλογος για 40 ονόματα για το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων. Και αυτά μιλάμε μετά από τι προκλήσεις του 2006 και θα συμπεριλάβει ο κατάλογο άλλα ονόματα ακόμη, ανάλογα με τι εξελίξει που θα υπάρχουν. Επιπροσθέτω, εξετάζουμε κάποιε επιλογέ για πιθανά μελλοντικά μέτρα που μπορούμε να λάβουμε και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ άλλων έχουμε καταστήσει σαφές ότι θέλουμε να συνεχίσουμε την ε, δέσμευσή μας, τη συνεργασία μας με την κοινότητα των πολιτών, με το λαό της Λευκορωσίας. Θα προχωρήσουμε με το θέμα της ε, χορήγησης ε, θεωρήσεων διαβατηρίου και θα έχουμε και τις σχετικές οδηγίες 28 Φεβρουαρίου εγκρίθηκε σχετική οδηγία. Ενθαρρύνουμε επίση τα κράτη-μέλη να ε, χρησιμοποιήσουν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τι δυνατότητε ευελιξία ε, του κώδικα για τι θεωρήσει διαβατηρίου, ιδίω ό,τι αφορά μείωση ε, των, του κόστου για την έκδοση μια θεώρηση διαβατηρίου. Επίση, έχουμε τετραπλασιάσει την παροχή βοήθεια προ την κοινωνία των πολιτών για το λαό τη Λευκορωσία. Παραμένουμε δεσμευμένοι υπέρ μιας ε, δέσμευση προ τη Λευκορωσία. Είχαμε και τα συμπεράσματα τον Ιανουάριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που τα επιβεβαιώνουν και ταυτόχρονα είναι σαφέ ότι οποιαδήποτε εμβάθυνση των διμερών μα σχέσεων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον θα έχει την βούληση η Λευκορωσία να τηρήσει τι αρχέ τη δημοκρατία του κράτους δικαίου και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αξιότιμοι βουλευτέ, θα ήθελα ολοκληρώνοντα να πω ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία παραμένει σε πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην μερίσια διάταξη της Κομισιόν και χαίρομαι που και το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει την πολύ σοβαρή συζήτηση και να μην ε, ε, επηρεαστεί από διάφορους περισπασμούς. Συνεργαζόμαστε στενά και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε εδώ η συζήτηση για τη Λευκορωσία, αγαπητοί συνάδελφοι, και μπορούμε να περάσουμε στι ψηφοφορίε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν καταρχά έξι προτάσει ψηφίσματο για τη Σρι Λάνκα. Μετά την έκθεση των ε, Ηνωμένων Εθνών, την παρακολούθηση της των Ηνωμένων Εθνών. Από ό,τι έχω καταλάβει,